Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια παρατήρηση διαδικαστική. Χθες, ενώ δεχτήκαμε μια αντιπροσωπεία από, τη από τους εκπροσώπους της Σιδηρουργίας στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Χαλιβουργίας, δύο συνάδελφοι δέχτηκαν επίθεση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι εργαζόμενοι ήρθαν για να συζητήσουμε το μέλλον τη ε, σιδηρουργία εδώ και τελικά τους περικύκλωσαν. Ήταν σαν συνωμοσία το που συνέβη. Ήθελα λοιπόν να το σημειώσω και χρειάστηκε να παρέμβουν ευρωβουλευτέ για να σταματήσει το επεισόδιο. Λοιπόν, ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να επιτρέπει στον καθένα την ελεύθερη έκφραση. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε να σας πληροφορήσω πως είναι γνωστά αυτά στον Πρόεδρο. Η διάσκεψη του Προέδρου, το Προέδρων θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα ε, βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Λυπούμαστε για το περιστατικό. Κάτι ακόμα επί της διαδικασίας, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να διαμαρτυρηθώ. Προετών ήμουν υπεύθυνο ε, για την έκθεση Κόρμπετ για να πάνε οι γραπτές ε, δηλώσεις από ένα γραφιάκι έξω από το ημικύκλιο. Και ήταν μια νίκη για την ε, δημοκρατία και τους απλούς βουλευτές. Ε, και τώρα η κυρία Ρατή, βοηθός Γενική Γραμματέας, το στείλε σε ένα απομακρυσμένο γραφιάκι. Παρακαλώ ξαναδείτε το γιατί είναι πλήγμα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία να μην είναι οι δηλώσεις εκεί που ήταν. Ευχαριστώ. Μάλιστα θα δούμε αυτά τα ζητήματα με την διάσκεψη των Πρόεδρων. Τελευταία δήλωση. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έγινε μία παρατήρηση από τον ε, σοσιαλιστή συνάδελφο για την ε, διαδήλωση των Χαλιβουργών. Ε, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μου διαπίστωσα με ντροπή πως έγιναν ζημίες σε κάποια δημόσια κτίρια και υποδομές του Στρασβούργου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Είπα από την αρχή πως θα δούμε το ζήτημα στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Τα περιστατικά είναι γνωστά και ο Πρόεδρος θα συζητήσει το τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρο ε, για αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε από την έκθεση Κάζα τώρα τις ψηφοφορίες. Τελευταία, δήλωση. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ένας από τους στόχου του Ευρωκοινοβουλίου είναι να προστατεύει τι μειονότητε. Θεωρώ ότι υπάρχει μειονότητα σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Εκείνη των καπνιστών. Πρέπει να υπάρξει ένας χώρος για κάπνισμα. Περνάμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ΚΑΖΑ. Υπάρχει ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. η έκθεση γίνεται δεκτή. Περνάμε στην έκθεση Φερέρα. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλές ονομαστικές ψηφοφορίες. Κύριε Πόσαλτ, ψήφισα αλλά δεν λειτουργήσε. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Μάλιστα, περνάμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Φερέιρα. Σημείο 1, το αρχικό κείμενο χωρίς τη ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε. Πέρας. Δεκτή. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 2 σε δύο μέρη. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο. Καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται περνάμε στο σημείο 6 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 15. Όχι ονομαστική. Διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο αρχικό κείμενο με δύο μέρη. Μέρος πρώτο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτή. Σημείο 10, τροπολογία 16, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε στο σημείο 11. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο. Σημείο 20 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Σημείο 21 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό σημείο 24 τροπολογία 17 τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές δεκτό περνάμε στο σημείο 24 τροπολογία 18 άρχεται η ψηφοφορία Ονομαστική. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 25 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή τροπολογία 20 επί του 26 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας Απορρίπτεται. Παραγραφός 33 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην παραγραφό 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δε... Απορρίπτεται. 39 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 1, μετά το εκτιμώντας α. Παρακαλώ, διανατάσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας γ, τροπολογία 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο. Διανατάσεως χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας G υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας J σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Εκτιμώντας κάπα σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Εκτιμώντας L με ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε τροπολογία 11 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας εν 12 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Εκτιμώντας τα τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Εκτιμώντας Y, ε, τροπολογία 14 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Εκτιμώντας ΑΒ υπέρ. Ε, Διανατάσεις χειρός παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας α δέλτα μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό νέο παράδειγμα Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Νέο παράδειγμα τροπολογία 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται. Ψηφίζουμε άρα το συνολικό κείμενο όπως έχει μεταβληθεί με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Η έκθεση εγκρίθηκε όπως έχει τροποποιηθεί. Περνάμε άρα στην επόμενη έκθεση. Παρακαλώ κυρία, κυρία εισηγητρία, κυρία Φερέιρα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική. Το θέμα είναι τι θέλει να πει το Ευρωκοινοβούλιο στο Συμβούλια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν καθορίζουν την οικονομική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2013, εγώ ε, έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περάσει ένα σωστό μήνυμα με ευρεία συνένεση. Όμω υπάρχουν διαφορετικέ πολιτικέ προτεραιότητε από τι διαφορετικέ ομάδε και αυτό ήταν σημαντικότερο τελικά από την ισχυρή και ενιαία θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Επειδή γνωρίζουμε μια κρίση άνευ προηγουμένου και εκρηκτικά ποσοστά ενεργεία στι περιφερειακέ χώρε τη Ευρώπη, θα έπρεπε εμείς ω ως εκλεγμένοι πρόσωποι, να είμαστε λιγότερο κομφορμιστές στην έκφρασή μα κατά τη λιτότητας. Μέτρα λιτότητας τα οποία επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αύξηση στη ζώνη ευρώ 0,7%. Αυτά δεν μπόρεσαν να περάσουν και έτσι επιτρέπουμε την συνέχιση ενός φαύλου κύκλου με καταστρεπτικές συνέπειες. Δεν συμφωνώ με αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι θα καταψηφίσω την ίδια την έκθεσή μου και δεν θα ήθελα το ε, όνομά μου να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των συντακτών της έκθεσης. Δεν στηρίζουμε τη συνέχιση αυτών των πολιτικών λιτότητα. ιδίως έτσι όπω εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και από ό,τι φαίνεται με τη στήριξη της πλειοψηφία των συναδέλφων αυτού του σώματος. Δεν εξυπηρετήσαμε σε τίποτα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η έκθεση εγκρίθηκε και περνάμε στην ψηφοφορία της επόμενης έκθεσης ε, της κυρίας Λόπε Φοντανιέ. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Παράγραφος 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Παράγραφό 17, μέρος πρώτο. Υπέρ. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Τα Αποχέ. Δεκτή. Τροπολογία 3 επί της παραγράφου 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται σημείο 29 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή παράγραφος 33 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. 36 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Τροπολογία 4. Διαματάσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Σημείο 42. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο διανατάσσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στο 42 τροπολογία 5. Παρακαλώ Διανατάσιο χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 Το αρχικό κειμένου σε δύο μέρη με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό το πρώτο μέρος. Μέρος δεύτερο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Παραγραφός 70, τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 76, αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ. Ε, με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 78. Το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μου λένε πως ε, η τροπολογία 7 είναι συμβατή με το άρθρο 76. Οπότε ψηφίζουμε και αυτήν. Η τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 78 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται εκτιμώντας α σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Εκτιμώντας H, με ονομαστική ψηφοφορία σε δύο μέρη υπέρ, ε, άρχιε ψηφοφορία του πρώτου μέρους. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Ναι, μέρος δεύτερο με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην υπολογία 9. Με ονομαστική ψηφοφορία. Έχει απορριφθεί το αίτημα για χωριστή ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στο παράρτημα σύσταση 5-2 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο, διανατάσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δέκτο. Σύσταση 7. Σε τρία μέρη. Και τα τρία με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτό. Μέρος τρίτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτό. Τροπολογία 10. Υπέρ. Διανατάσεως χειρός. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο συνολικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και γίνεται δεκτό. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Με συγχωρείτε επί τη διαδικασία. Κυρία συνάδελφε. Έχετε το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να πω με συντομία στους αδέλφους της δεξιάς ότι τώρα ψηφίσανε κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση 100% με την προηγούμενη έκθεση που ψηφίσανε. Για βάλτε τη μία έκθεση δίπλα στην άλλη και συνειδητοποιήστε τι έγινε. Παρακαλώ να μείνετε επί της διαδικασίας. Αυτό δεν ήταν επί της διαδικασίας. Περνάμε στην τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά αποχές δεκτό τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία απορρίπτεται ε, με συγχωρείτε πέρας απορρίπτεται Περνάμε στην τροπολογία 6 δέλτα, δυνατά στους χειρός υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο εκτιμώντας α ν σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας AQ σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας ΑΛΦΑ τάφ σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε γιατί δεν είναι σίγουρο άρχεται η ψηφοφορία πέρας δέκτο μέρος δεύτερο διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο εκτιμώντας AV. Μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας ε σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας ζ υπέρ κατά αποχές δεκτό μετά το 10 τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε άρα το κείμενο όπως τροποποιήθηκε χρειάζεται η ειδική πλειοψηφία 378. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στο ψήφισμα για κατεξουσιοδότηση κανονισμό, κανονισμούς της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο. Κυρία Επίτροπε. Ε, Στις 4 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ένα ψήφισμα και απέρριψε δύο από αυτές τις κατανάθεση πράξεις σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που συμπληρώνουν τον 648 2012 σε σχέση με αυτά τα παράγωγα και σε σχέση με αυτά τα εμπορικά καταπιστεύματα. Οπότε θα πρέπει προσεκτικά να εξετάσουμε τους λόγους αυτή της απορρίψεως, διότι εμείς στον βωμό συμβιβασμού πρώτη να εξασφαλίσουμε το ότι όταν γίνει η, έντυση, η, ε, γίνει η έγκριση για αυτά τα χρηματιστηριακά προϊόντα και οπότε θα, πρέπει να γίνει αυτή η εγκαθάριση από, αυτού του αυτούς τους φορείς τα τάξη χρηματιστηριακά παράγοντα, του κεντρικού αντισυμβολόμου και τα αρχεία. Οπότε και εμεί συμφωνούμε ε, με το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της ασφαλείας του δικαίου και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προβεί στην ακόλουθη δήλωση. Απεφασίσαμε το ότι αυτού του είδους οι προδιαγραφές θα πρέπει να βασίζονται ε, στο σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών που προετοίμασε η ΕΣΜΑ. Οπότε είναι δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη να εξασφαλίσουμε το ότι όλοι αυτοί οι κίνδυνοι θα υπόκεινται σε εποπτεία, θα τη θα και έτσι θα προστατεύεται η οικονομία. Αντιλαμβανόμεθα που έγινε η επιφυλάξη σα. Οπότε πρώτη θέμεθα να διασφαλίσουμε το ότι όταν αυτή η απόφαση εγκριθεί όσον αφορά αυτού του είδους τα παράγωγα, τα εξωχρηματιστηριακά, τότε οι υποχρεώσεις από μη χρηματιστηριακές ε, εταιρείε να κάνουν την εκαθάριση πρόκειται να είναι καθορισμένες με ακρίβεια και θα υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες και περίοδοι όπως προτείνονται για τις τραπεζικές εγγύησεις. Οπότε αυτές οι εταιρείε θα έχουν αρκετό χρόνο να προσαρμοστούν στο νέο τοπίο. Ταυτόχρονα έτσι θα έχουμε κάποια ε, λογική προσέγγιση. Και σχετικά με την EMA θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο α του ίμια πρόκειται να ισχύσει στο μέλλον. Και επομένω, η ανάπτυξη αυτών των τεχνικών προδιαγραφών είναι κάτι που αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και είμαι θα βέβαιη ότι αυτή η διαδικασία πρόκειται να προσαρμοστεί και να τελειοποιηθεί στο μέλλον. Οπότε χέρι-χέρι με το κοινοφούλιο και με ανοιχτό διάλογο και διαφάνεια πρόκειται να προχωρήσουμε για αυτά τις τεχνικές προδιαγραφές. Όμως να υπάρχει και αρκετό χρονικό διάστημα για να κινηθούμε και ε, να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε στα πλαίσια της διοργανικής συμφωνίας, συγκεκριμένα δε όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των κατεξιοδότηση πράξεων και σε σχέση με την ανάπτυξη των ε, καλών πρακτικών πρόκειται να προωθήσουμε αγαστές ε, δημιουργικές σχέσεις με τακτές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ημών και ημών όσον αφορά αυτές τις προδιαγραφές και θα λάβουμε υπόψη ό,τι έχει συμφωνηθεί διοργανικά σε σχέση με το πώς θα καταλήξουμε να συμφωνήσουμε για αυτές τις κατοξιώδεις πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στην πρόεδρο της ε, Αρμόδιας Επιτροπής, την κυρία Σάνου Μπούλς αντιμετωπίσαμε προγράμματα, προβλήματα συγγνώμη, με αυτά τα τεχνικές προβλήματα της MEA και όσον αφορά ε, το, το, περιεχόμενο, όσον αφορά τη συνεργασία και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ε, και βεβαίω θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεσμεύθηκε επ' αυτού και διότι προέβη σε αυτήν την ε, δήλωση ε, οπότε τώρα προτίθενται να αντιμετωπίσουν, να επιλύσουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει. Επίσης δε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διαβεβαιώσει ότι πρόκειται να γίνουν βήματα προ το μέλλον, βήματα προόδου με καλύτερη συνεργασία όσον αφορά τα διαδικαστικά. Επίση σα διαβεβαιώ ότι όσον αφορά κάποια από τα προβλήματα με, το χρονοδιάγραμμα, ήδη σήμερα έχουμε αναλάβει τα διαβήματα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερε διασφαλίσει όσον αφορά το κείμενο του πρώτου επίπεδου. Οπότε, ε, βεβαίω τώρα αυτό είναι, είναι παρθένο, είναι νέα, νέα περιοχή, νέα πράγματα. Ε, αλλά θα συνεχίσουμε να προωθούμε το κείμενο και επίσης ευχαριστούμε για αυτές τις διαβεβαιώσεις ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα ε, και θα πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε τακτή επαφή μαζί μας, θα υπάρξουν ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά επίσης προσδοκούμε να υπάρξει μια συνέχεια όσον αυτά τα τροποποιημένα τεχνικά ζητήματα και προδιαγραφές ε, ε, ε, το χρόνο και επομένω σα ευχαριστούμε και ε, εκ μέρου του κ. Λάγκεν και εκ μέρου τη Οικονομική μας Επιτροπής. Ευχαριστούμε ε, και πρόκειται να γίνει ακριβώ η απόσυρση αυτή του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Οπότε δεν ψηφίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα, δηλαδή το ψήφισμα για την 22η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία πέρας δεκτή. Σημείο 62 σε δύο μέρη. Εδώ πέρα η συγγήτρια θέλει να καταθέσει μια προφορική τροπολογία. Κυρία Αντρικένε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητήσαμε να γίνει κατά δύο στην παράγραφο 62. Θα ήθελα να σας προτείνω μια προφορική τροπολογία όσον αφορά αυτήν την ε, τροπολογία εις δύο τμήματα. Πρώτον, προσθέτουν και να ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεύτερο τμήμα όποτε είναι δυνατόν. Παράγραφος 62 επομένω, εάν τροποποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα έχει ω εξή. Προσδοκούμε την ανάπτυξη στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συντονιστούμε με τι δράσει του ΟΗΕ και των φόρουμ του ΟΗΕ. Και επίση διατυπώνεται η σύσταση για, με Υπάρχουν επικοινωνίε στρατηγικές προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιούνται όποτε είναι δυνατόν, ούτω ώστε να προβάλλεται το πόσο για όλε αυτέ τι χώρε έχει δεσμευτεί και στρατευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένως ε, να υπάρξει υποστήριξη για αυτή την πολιτική. Ε, δεν χρειάζεται κατά διέλευση ψηφοφορία εάν το κείμενο εγκριθεί όπω σα το διάβασα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Έχει κάποιο αντίρρηση για την προφορική αυτή τροπολογία. Εάν όχι, περνάμε σε ψηφοφορία σε ένα μέρος του αρχικού κειμένου όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Περνάμε στην τροπολογία του συνολικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο ψήφισμα για την δικαστική εκπαίδευση και τους δικαστικούς συντονιστές. Δεν έχουμε καμία τροπολογία. Υπέρ του ψηφίσματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην έκθεση Μάουρο. Μία τροπολογία έχω. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε το συνολικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ. Μια που τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους που δεν θέλουν να κάνουν επεξηγήσεις ψήφου, να εγκαταλείψουν την αίθουσα γρήγορα, έτσι ώστε να περάσουμε αμέσως στις επεξηγήσεις ψήφου.